να υποβάλλετε τις προτάσεις σας και αυτό έχει συμφωνηθεί με όλες τις πολιτικές ομάδες. Η συζήτηση για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο χώρο του Σέγγεν θα περιλάβει και ε, προφορικές ερωτήσεις από τους φιλελεύθερους, την Ηνωμένη Αριστερά και ε, τους Ευρωπαίους Ομοσπονδιακούς Δημοκράτες. Όσον αφορά την κατάσταση ε, για την, για την Ιεμένη ε, ε, και τον Μπαχρέιν θα διευρυνθεί και θα περιλαμβάνει και την Συρία και την Αίγυπτο και επιπλέον μία δήλωση του αντιπροέδρου, της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της προσώπου για τις εξελίξεις στην Ουκρανία θα περιληφθεί στη συζήτηση με την Ιεμένη, Μπαχρέιν, Συρία και Αίγυπτο ε, το ψήφισμα θα ψηφιστεί στην δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Όσον αφορά τις ομιλίες ενός λεπτού, αυτές ε, θα ληφθούν αμέσως μετά τη συζήτηση για την Ουκρανία και τέλος η συνεδρίαση θα επεκταθεί μέχρι τις 10 ε, το βράδυ. Τώρα, όσον αφορά την Πέμπτη, η έκθεση της κυρίας Σάρον Μπολ σχετικά με τον καθορισμό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης θα περιληφθεί εις ε, ε, τον χρόνο ψηφοφοριών και δεν υπάρχει προθεσμία για τροπολογίες. Έχετε κάποια αντίρρηση, σχόλια, δεν βλέπω κανένα. Οπότε έτσι προχωράμε σε ε, μία πρόταση η οποία έχει προβεθεί αλλά βλέπω ο κύριος Γκολνής ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω να κάνω μία παρατήρηση σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση που προβλέπει μία συζήτηση για την κατάσταση στην Ιεμέρη και στο Μπαχρέιν που επεξετάθη στη Συρία και στην Αίγυπτο. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά αλλά είναι κράτη τα οποία δεν επηρεάζουμε άμεσα. Ενώ, ενώ ο Ευρωπαϊκός στρατός μαζί με τον ΟΗΕ συνεχίζει και μαζί με το ΝΑΤΟ να ε, σκοτώνει τους ε, αντιτιθέμενους στο τονό καθεστώς στην ε, Λιβύη και στην Σύρτη. Πρόκειται για πάρα πολλούς νεκρούς και δεν πρέπει απλώς να ακολουθούμε τις επιταγές του ΝΑΤΟ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Τώρα έχω, έχουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, σε ό,τι αφορά την κατάθεση ψηφισμάτων σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την κατάσταση στην Ιεμένη, τον Παχρέιν, τη Συρία και την Αίγυπτο και τη σχετική προθεσμία. Το ΕΛΚΑ ζήτησε